So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Heute Morgen zu unserer Σας καλωσορίζω στη σημερινή μα συνεδρίαση με μία σειρά ψηφοφοριών Βρισκόμαστε στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης. Εξουσία ανάθεση νομοθετικού έργου. Και αυτή είναι μια γνωμοδότηση που έχω προετοιμάσει εγώ ίδιο για την ορτή νομικών υποθέσεων στην έκθεση Σάιερ. όσον αφορά την ε, ανάθεση εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν 14 τροπολογίες. Έχετε όλες σας τις κάρτες ψηφοφορία μαζί σα, γιατί αν υπάρχουν ασάφειες θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά αν δεν την έχετε μαζί σας, παρακαλώ φροντίστε να την αποκτήσετε. Αρχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία του σημείου 10. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εντάξει, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Θα ελέγξουμε συχνά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Το ΕΛΚ έχει τρεις παραπάνω. Ας φροντίσει ο συντονιστής. Κανένας δεν έχει περιτούς, ε. ε. Καλά θα ήταν να έχουμε πιο πολλούς. S&D is eine zu Σοσιαλιστές ένας παραπάνω. EVP immer Το ΕΛΚ θα ακολουθεί να έχει δύο περισσότερους από ό,τι χρειάζεται. Σοσιαλιστές έναν περισσότερο. ΕΚ ακόμα έναν και οι σοσιαλιστές έναν. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα περισσότερο από ό,τι πρέπει. Ωραία. Τώρα εντάξει, πέρασε η ψηφοφορία. 39 υπέρ, 21 κατά, όπως τους είδα. Ε, εγκρίθηκε δηλαδή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Με μια προφορική τροπολογία της κυρίας Άση. Ποιος είναι υπέρ της τροποποιημένης τροπολογίας. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7.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 PPE hat immer noch... Το έλεγχο εξακολουθεί να έχει δύο περισσότερους από ό,τι πρέπει. Έναν ακόμα. Ένα ακόμα περισσότερο από ό,τι πρέπει στο ΕΛΚ. Ωραία. Τώρα εντάξει. 33 υπέρ 28 κατά. Είναι κρίθη. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχισε ψηφοφορία. Το έργο έχει πάντα έναν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Για να οργανωθείτε καλύτερα παρακαλώ. Να μην χρειάζεται να το λέω συνεχώς. Ωραία. Λοιπόν, 62 είπε, κανένας κατά, ευχαριστώ πολύ. Πέρα τη ψηφοφορία. Ε, γίνεται δεκτή η γνωμοδότησή μα. Ωραία. Και τώρα. Ja. Yeah. Wir kommen zu dem spannenden Punkt 11. Λοιπόν, περνάμε στο πολύ ενδιαφέρον σημείο 11 τη ημερησία διάταξης. Παροχή πληροφοριών για το τρόφιμα στου καταναλωτέ. Έκθεση Ρενάτε Ζόμερ. Διαδικαστικά κυρία Ζόμερ, εισαγωγικά. Να, με κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι για το τεράστιο αυτό θέμα. Προετοιμάσαμε την ε, τον κατάλογο ε, ψηφοφορία χθε το απόγευμα. 73 σελίδε, 900 τροπολογίε περίπου. Υπήρχε μια ε, προθεσμία την περασμένη Παρασκευή στι 11 το μεσημέρι για συμβασικέ ψηφοφορίε, παγιωμένε κλπ. Και κατά τμήματα ψηφοφορίε. Αυτή η προθεσμία δεν ελήφθη υπόψη. Μέχρι τελευταία στιγμή υποβλήθησαν προτάσει, ιδίω για κατά τμήματα ψηφοφορίε που την υπόψη. Εκτό αυτού, χθε το μεσημέρι μόλι ενημερώθηκα από τη γραμματεία, χωρίς να έχω ενημερωθεί, ότι έχουν συμπεριληφθεί τώρα δύο παγιωμένε ε, ε οι οποίε ανατρέπουν όλο το κατάλογο ψηφοφορία και εγώ δεν ε, μπόρεσα λόγω του περιορισμένου του χρόνου να ελέγξω κατά πόσον αυτά ήταν σωστά πια. Οι αναφορέ ε, στον κατάλογο ψηφοφορία δεν μπορούσα να τις λέξω ότι μπορούσα να προσαρμόσω τις δικές μας συστάσεις για ψηφοφορία. Και χθες το βράδυ είχαμε μια συζήτηση με τους συναδέλφους χωρίς ε, τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ο θυμός ήταν τεράστιος, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε έτσι χωρίς ένα τόσο τεράστιο θέμα. Γιατί είχε λήξει η προθεσμία και μέχρι τη στιγμή στιγμή τροποποιεί το, ο τη ψηφοφορίας χωρί να ενημερωθώ, χωρί να έχω το χρόνο να την εξετάσω, και γι' αυτό δεν μπορούσα να, ε, ε, να τηρήσω τις υποχρεώσεις μου ως ε, ε η Γι' Αυτό προτείνω να βληθεί η ψηφοφορία στην επόμενη μας συνεδρίαση. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Σόμερ. 900 τροπολογίες. Πραγματικά είναι μια έκτακτη πάντα κατάσταση, πολύ δύσκολη για όλους, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, Έχω να πω ως πρόεδρος ότι ο κατάλογος ήταν γνωστός εδώ και 15 μέρες. Οι ομάδες ενημερώθηκαν την περασμένα Τρίτη στο Στρασβούργο για τον κατάλογο ψηφοφορίας και του συζητήθη η τοποθέτησή τους μέχρι την Παρασκευή. Διοικητικά είχαμε πει μέχρι την Παρασκευή στις 11 το μεσημέρι να έχουν ληφθεί υπόψη όλες τις τροπολογίες κλπ. Αλλά αν κοιτάξετε το κανονισμό μας βλέπετε ότι μπορούν να υποβληθούν ε, αιτήσει για κατημήματα ψηφοφορίες μέχρι την παραμονή μιας ε, ψηφοφορία. και είναι πολύ λίγε. Για από τις 900 τροπολογίε, πολύ λίγε είναι αυτέ. Και όσον αφορά τι συμβαστικέ τροπολογίε, πρέπει πάντα να ρωτήσω κατά πόσον συμφωνεί η ολομέλεια τη επιτροπή μα. Μπορεί κανένα να πει και όχι, αν έχει αλλάξει κάτι. Και βέβαια για τις συμβιβαστικές τροπολογίες πάντα είμαστε έτσι γενναιόδοροι και λέμε ότι αν μπορούν να συνενωθούν διάφορες τροπολογίες ας ψηφίσουμε όχι τυπικά αλλά επί της ουσίας. Και για μένα ήταν δύσκολα τα πράγματα, ομολογώ, να εξετάσω αυτό τον πίνακα. Τυπικά έχω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψηφίσουμε σήμερα. Εάν υπάρχουν διαφωνίες, ζητήσατε εσείς ε, να αναβληθεί, μπορούμε να ψηφίσουμε από αυτό. Ας το κάνουμε όπως είναι Ολμέλεια, να μιλήσει ένας υπέρ και ένας κατά. Ο Πέτερ Λίζε υπέρ και κάποιος θα μιλήσει κατά. Η Λίνα Μακέβεν κατά. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα κατά πόσο νομικά τυπικά είναι σωστό ή όχι δεν μπορούμε να το εξετάσουμε αυτή τη στιγμή στα γλίγορα. Μπορεί να αποφασίσει ο πρόεδρος, θεωρώ. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει οπωσδήποτε αν δεν έχουμε τόσο μακρά συνεδρίαση να τροποποιήσουμε τη διαδικασία. Γιατί υπήρχε το πρόβλημα για όλες τις πολιτικές ομάδες ότι χθε δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε το σύνολο της ομάδας ψηφοφορία. Γιατί βέβαια είναι διαφορετικό κατά αν έχω μια προσωρινή λίστα ψηφοφορία ή κατά θα έχει λίγη, Γιατί μία και μόνη τροπολογία μπορεί να αλλάξει την ψηφοφορία για ένα ολόκληρο άρθρο. Γιατί αν αλλάξει η σειρά των τροπολογιών θα πρέπει να σκεφτώ κατά πόσον εκεί θα βάλω μείον αντισύν γιατί η δική μας τροπολογία θα καταπέσει κλπ. Αυτό το κάνουμε συνεχώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι ίσως τυπικά είναι σωστό ότι υπήρχε αυτός ο κατάλογος πριν από δύο εβδομάδες, αλλά τελικός κατάλογος ψηφοφορίας προετοιμάστηκε χθε το βράδυ στις 5. Και αυτό οπωσδήποτε ήταν προβληματικό για όλες τις πολιτικές ομάδες. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σημειωθεί το νομικό θέμα, να το ξαναεξετάσουμε. Αλλά το πώς θα εργαστούμε την επόμενη φορά θα ήθελα να πω ότι να συζητηθεί στους συντονιστές. Δηλαδή να δοθεί επαρκής χρόνος πριν από ψηφοφορία σε όλους να εξετάσουν μια ένα τελικό κατάλογο ψηφοφορίας. Και αυτό επειδή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, χωρίς να κατηγορήσω κανένα. Γιατί αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη έκθεση στην Επιτροπή μας, όλοι είχαν προβλήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος έσφαλε, αλλά η κατάσταση που δημιουργήθηκε ίσως θα οδηγήσει σε σφάλματα να ψηφίσουμε τώρα. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω με όλη την καλή βούληση να αναβάλουμε την ψηφοφορία αυτή δεν ε, πειράζει γιατί εδώ και 18 μήνες έχουμε την πρόταση Κομισιόν επιτάπτως. Άμα την αναβάλουμε για άλλο ένα μήνα δεν πειράζει και θα μπορούσαμε τότε να πούμε ναι, ξέραμε ακριβώς τι ψηφίζαμε και δεν το ξέρουμε σήμερα και αυτό παρακαλώ να ακολουθήσετε την πρόταση της συζητήτρες. Ωραία, λέει ο Ακούσαμε εκείνους που ήταν υπέρ. Η Λίντα κατά τώρα. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα το θέμα. Αυτό μας απασχολεί μακρόν στο Κοινοβούλιο και γνωρίζουμε το όλο θέμα. Βεβαίως τον κατάλογο ψηφοφοριών τον λάβαμε χτες, αλλά γνωρίζαμε το προσχέδιο, τα, οι τροπολογίες είχαν υποβλήθει, ξέραμε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν υπηρετούμε κανένα με μία αναβολή η κυρία Γουίλμοντ, η Σκιώδη, ζήτησε από, τον εισηγητή, από την εισηγήτρια να ε, αναβάλει την ψηφοφορία και τότε είπε ότι όχι, γιατί ε, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν ε, τροπολογίες συμβιβασμού, αλλά παγιωμένες. Γι' αυτό χθες η εισηγήτρια δεν είπε τίποτα τέτοιο περί αναβολής. Εμείς περάσαμε πολλές ώρες χτες το βράδυ, είδαμε τον κατάλογο και πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Γνωρίζουμε τα θέματα, ξέρουμε ποιες είναι οι διαφορές και ποια ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Yeah, ναι, είναι αυτό μόνο βέβαια. Η Επιτροπή μας μπορεί να αποφασίσει, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Όποιος είναι υπέρ της αναβολής,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 Λοιπόν, το ΕΛΚ έχει κάποιους παραπάνω. Ακόμα, οι σοσιαλιστές το ίδιο. Βέα, Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Πέρες πληροφορίες. 21 υπέρ 30 κατά της αναβολής. Με μία αποχή. Der Απορρίπτεται λοιπόν η πρόταση της ηγετρίας. Η Ηγετρία; Πρόεδρε. Απερίφθη η πρόταση. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά αμφιβάλλω κατά πόσον εμείς ε, σαν επιτροπή μπορούμε πραγματικά να δώσουμε τη τελική μας άποψη και παρακαλώ οι επιφυλάξει να συμπεριληφθούν στα πρακτικά και θεωρώ ότι οι υπηρεσίε θα εξετάσουν το νόμο της ψηφοφορίας που θα πραγματοποιήσουμε τώρα να το εξετάσουν λέω και, ελπίζω, και παρακαλώ και η διάσκεψη του Προέδρου να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πρόεδρος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξεταστεί οτιδήποτε. Όπως σας είπα, υπευλήθησαν κατά τμήματα ψηφοφορίας αργότερα και αυτό είναι ε, επιτρεπτό σύμφωνα με τον κανονισμό. Υπάρχουν δύο παγιωμένες ε, ε, τροπολογίες, μπορεί κανένας να κατεψηφίσει. Τυπικά δεν υπάρχει σφάλμα λοιπόν. Δεν ξέρω τι πρέπει να εξεταστεί δηλαδή. Υπάρχει μια δέσμη 900 τροπολογιών εδώ και 18 μήνες το ξέρουμε το θέμα. Λοιπόν, ωραία. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία πρέπει να εξετάσουμε και ένα άλλο θέμα. Το κατά πόσον πολλές από τις τροπολογίες είναι 162 της κυρία Ζόμερ για το προφίλ του Ευρωπαϊκού 525 της κυρία Ζώνα για την ε, Διαχειριστική Επιτροπή της Υπηρεσίας 526 ε, του συναδέλφου Σλούτερ για την αλλαγή της κοινή οργάνωσης αγοράς για τα προϊόντα αλίας και ε, ηχθειοκαλλιέργειας και τροπολογίες για την σήμανση των των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων 224, 361 και 511. Εκτός από την 526 του κυρίου Σλούτερ, οι άλλες ε, τροπολογίες σχετίζονται με την ψηφοφορία μας. Και εγώ ως πρόεδρος αποφασίζω ότι θα ε, είναι επιτροπή η, ψηφοφορία από αυτόν. Η 526 όχι, γιατί η κοινή οργάνωση αγοράς και η προστασία των αριθμητικών αποθεμάτων δεν είναι θέμα που μας αφορά εδώ, που μας αφορά η ενημέρωση των καταναλωτών για το περιεχόμενο των τροφίμων. Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναγκασμένα την κάνουμε. Αλλά η Επιτροπή μας ήδη στο REACH ε, κατάφερε ακόμα περισσότερα και θα φροντίσουμε να τα καταφέρουμε και εδώ. Λοιπόν, τροπολογία 34. Υπέρ, κατά αποχές για να δούμε καλύτερα ηλεκτρονικός έλεγχος Ein EVP zu viel. Könnten die Koordinatoren nicht δεν μπορούν οι συντονιστέ να δουν τώρα ποιο ψηφίζει και ποιο δεν ψηφίζει, γιατί μου φτάνει. Genommen 33 gegen 26. Bei einer Enthaltung. Λοιπόν, 33 υπέρ 26 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος.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 Πείτε, Λίζα, ρίχα σε μάμπου, δεν μπορείτε να μετρήσετε. Immer noch einer. Eine oder einer. Ja, kann einer dafür sorgen, dass es... Μήπως μπορεί κάποιος να φροντίσει ε, να είναι ο σωστός αριθμός των μελών. Λοιπόν, εντάξει, 29 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. 36. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 15 υπέρ. Κατά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 κατά αποχές μάλλον έγινε δεκτή αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικός έλεγχος Abstimmung geschlossen. Πέρας 32 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 και 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι επόμενες καταπέφτουν 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αγκρί 18 υπέρ κατά Εποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 19. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Άρχιτη ψηφοφορία. Εξακολουθεί να υπάρχει ένας περισσότερος από ό,τι πρέπει στο ΕΛΚ. Τώρα είμαστε εντάξει. 24 υπέρ 35 κατά. Απερίφθη. Παρακαλώ. Συνάρθω Δούτσκι. Ευχαριστώ το μηχάνημά μου για την ψηφορία δεν λειτουργεί. Κάποιο μπορεί να με βοηθήσει, ίσω. Ένα τεχνικό. Ναι, ναι, θα έρθει αμέσω. Για να μπορεί και ο να ψηφίζει ηλεκτρονικά. Ωραία. Wo weiter? 256. 256 καταπίπτει. 257 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Να ελέγξουμε. Μάλλον έγινε δεκτή, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Abstimmung geschlossen. Πέρα ψηφοφορίες. 32 υπέρ, 27 κατά. Ενεκρίθη. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 και αγκρή 20. Ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 53. Abstimmung beendet. Ja, 32. 32 υπέρ, 29 κατά εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 258 υπέρ. Α, όχι. Α, συμβατή, ναι, ναι. Ήμκο 18. Στο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 258. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 260 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 262 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 263 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εξήντα Υπέρ της 61. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε 62. Άρχη ψηφοφορία. Abstimmung geschlossen. ψηφοφορία. Ναι, 32 υπέρ, 27 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Άγκρι 24. Η 63 είναι γλωσσική φύσεω και μετά περνάμε στην 268. Με ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτη τμήμα, παρακαλώ, υπέρ. Dagegen Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε. Αυτή ήταν η άγκρη 24 και 268. Περνάμε τώρα στην 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, τροπολογία, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την ΙΜΚΟ 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την ΙΜΚΟ 22 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Abstimmung beendet. Ja, habe ich richtig gesehen. Μάλιστα, καλά τα είδα. Λοιπόν, 32 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. Για την 68. Καταπίπτει. Και περνάμε στην 69 παρακαλώ. Για την 69 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 71. Wer ist für 71? 71 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Kommen wir zu 275. Περνάμε στην 275 με προφορική τροπολογία. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Beendet. Πέρασα. Ήταν πραγματικά δύσκολο να το δω. 30 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται ως εκ τούτου. Και περνάμε στην 72. Α, συγγνώμη. Έχουμε ψηφίσει την προφορική τροπολογία η οποία και απορρίφθηκε. Τώρα θα ψηφίσουμε όμως και την 275 όπως είχε στο αρχικό κείμενο. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Βλέπω ακριβώς την ίδια σύνθεση. Απορρίπτεται, αλλά άμα θέλετε να το ελέγξουμε, το ελέγχουμε ωραία. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Α, κοίταχτε που κάτι άλλαξε. Κάποιος άλλαξε γνώμη. 29 υπέρ, 31 α, κατά, απορρίπτεται όπως και πριν. Περνάμε τώρα στην 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 278 καταπίπτει και έτσι περνάμε στην άκρη 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άκρη 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Because we adopted λέει ο πρόεδρος, επειδή αγκρίναμε την 59. Και γι' αυτό λοιπόν καταπίπτει. Το βλέπετε στα σχόλια, στις παρατηρήσεις. Το 74 zurückgezogen, 75 dafür. 75 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Και τώρα Περνάμε στην 280 και στην ΕΜΚΟ 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 281 281, παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Για την 283 λέει ο πρόεδρος. Beendet. Πέρας Είναι σαφές το αποτέλεσμα. 39 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει πίπτη 25 ή 67, 76 παρακαλώ. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 285. 282. 285. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι σαφές το αποτέλεσμα, αλλά ας το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας για την 285 παρακαλώ. Πέρας. Είναι σαφέ το αποτέλεσμα, σαφέστατο. 77. Ακόμα θα λειτουργεί η συσκευή σα. Όχι, ναι, ευχαριστώ. Απλά να εξηγήσω το εξή. Από ό,τι κατάλαβα, αποδεχτήκαμε, εγκρίναμε την 76 και τώρα αναφέρεται στο αρχείο μου ότι καταπίπτει 282 αν ευκριθεί 76, σωστά. Μα δεν ψηφίσαμε την 282, την 285 ψηφίσαμε. Sorry. So it's mistaken in, in a... Άρα είναι λάθος. 77 παρακαλώ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν και περνάμε στην 28 υπέρ.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 Εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτονται. Ας το ελέγξουμε. Έναρξη παρακαλώ ψηφοφορίας. Πέρας. Οριακό το αποτέλεσμα, αλλά απορρίπτηκαν. απορρίφθηκαν. Άγκρι 28, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 289 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Οριακό το αποτέλεσμα πρέπει να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας για την 289. Πέρας. Good. Απορρίπτεται 29 υπέρ, 32 κατά, 290 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 και ΙΜΚΟ 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγρι 29 και 292 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΜΚΟ 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Περνάμε στην 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμικο 32 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 32. Υπέρ. Κατά. Θέλω να πω ένταξη ψηφοφορίας. Πέρας. 32 ψήφι. υπέρ, 30 κατά, εγκρίνεται. Ήμκο 32, λέει ο πρόεδρος υπέρ. Αυτή ψηφίσαμε. Εντάξει. 295 και 297 και η άγκρη 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην ενοποιημένη τροπολογία υπερθμών 2 με με ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά του πρώτου τμήματος παρακαλώ. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι μάλλον θετικό το αποτέλεσμα, αλλά ένα ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά να το ελέγξουμε. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Εντάξει ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 32 ψήφοι υπέρ, 29 κατά μία αποχή εγκρίνεται. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι ίδιο είναι το αποτέλεσμα, αλλά ας το ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Εντάξει ψηφοφορίας. Πέρας. 33 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Και συνεχίζουμε στη σελίδα 12. Κάτω-κάτω στην 316. 316 ψηφίζουμε. 316. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Και περνάμε στη σελίδα 13 τώρα, στην 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90, Άγκρι 33, Ήμκο 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 318 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 319 ΙΜΚΟ 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, ήταν σαφές το αποτέλεσμα, αλλά αν θέλετε το ελέγχουμε. Ποιος θέλει έλεγχο. Εντάξει, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρακαλώ. Πέρας. Ήταν σαφέστατο το αποτέλεσμα. Καταπίπτει η άγκρη 35, περνάμε στην ύμικο 36, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Άγκρη 36, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 92, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 93 και ύμικο 37, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 320 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και περνάμε έτσι στην ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι η ενοποιημένη τροπολογία υπεριθμών 3 καταπίπτει. Και συνεχίζουμε στη σελίδα 15. Στην ενοποιημένη τροπολογία υπεριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στη σελίδα 16 η 331 και η ΙΜΚΟ 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98, 42, 335 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98, άγκρι 42 και 335 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συνεχίζουμε. Η 334. Ψηφίζουμε υπέρ. Για την 334. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικής παρακαλώ. Τώρα περισσεύει ένας από τους σοσιαλιστές. Ακόμα. Από τους σοσιαλιστές παρακαλώ ένας να βγάλει την κάρτα του. Εξακολουθεί να περισσεύει ένας από τους σοσιαλιστές. Πρόεδρε. Λέει εδώ ότι, ότι η 4 κατα πίπτει εάν η 98 εγκριθεί και από όσο βλέπω, από όσο ξέρω, έχει εγκριθεί η 98. Έχετε δίκιο. Άρα δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε το σημείο αυτό εφόσον εγκρίθηκε η άγκρη 42, καταπίπτει η 334 και το ίδιο ισχύει και για τις επόμενες, το επόμενο σημείο. Και άρα συνεχίζουμε. Ήμκο 44. Στη σελίδα, ε, στην επόμενη σελίδα, ΙΜΚΟ 44. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 43 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας κάτι να, κάνει, να κάνουν οι σοσιαλιστές γιατί εξακολουθεί να περισσεύει ένας τώρα μάλιστα, εντάξει, ή όχι. Είμαι Όχι, έχουμε ακόμα έναν παραπάνω. Τώρα εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. Σωστά το είχα δει, 31 ε, υπέρ, 30 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. 3.41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 και άγκρι 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 343. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 344. Άγκρι 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε για την 3.47 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 35, 25, υπέρ, 25 κατά, εγκρίνεται, ναι. 101. Α, συγγνώμη, η 100. Η 100 παρακαλώ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε για την 101. Έναρξη ψηφοφορίας. Περισσεύει ένας από τους σοσιαλιστές. Εντάξει. 35 υπέρ, 26 κατά. Εγκρίνεται. Τρία σαράντα εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμικο 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Στην 350 θα ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Επειδή το πρώτο τμήμα είναι ταυτόσιμο με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα δεν χρειάζεται τροποποίηση, τροπολογία. Για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έγινε κάποιο λάθος. Αν κοιτάξετε το κατάλογο ψηφοφορία, κάτω από το δεύτερο τμήμα αναφέρεται ότι καταπίπτει αν, αν εγκριθούν τροπολογία 1 ή 2 ή αν... Ε- Α, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει η κυρία Ζόμερα, εγώ έκανα λάθος. Ναι, το είδατε, το είδατε. Ότι εσείς κάνετε λάθος και γι' αυτό λοιπόν διαγράφει. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα και περνάμε τώρα στην 103. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 351 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι ήταν σαφές το αποτέλεσμα, αλλά αν θέλετε ας το ελέγξουμε για την 353 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Σαφές το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε φτάσει στην άγκρη 50 και στην 352. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η επόμενη και η μεθεπόμενη. Και συνεχίζουμε στην 357 του κυρίου Σλίτερ. 357 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107-356 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 359 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 360 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας για την 360. Abstimmung Πέρας. 35 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ η κυρία Ζόμαρ ναι θα ήθελα να αποσύρω την 110 αποσύρθηκε λοιπόν από την κυρία Ζόμαρ ευχαριστώ Άγκρι 51 σχόλιο εκτός μικροφώνου ότι εγώ θέλω να συμπεριληφθεί. Αν θέλει λοιπόν κάποιος να συμπεριληφθεί θα πρέπει να την ψηφίσουμε. 110. Ποιος είναι υπέρ της 110 παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. Όχι, είναι σαφές το αποτέλεσμα, σας παρακαλώ, ότι είναι σαφές. Αλλά εφόσον απαιτείται έλεγχο, ας το ελέγξουμε. Πέρας ψηφορίας. 37 ε, ψήφοι υπέρ, 22 κατά, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άγκρι 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 361. Κάρλ Σλίτερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 362 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Γιατί έχετε... Δεν σηκώνετε και τα χέρια σας και δεν μπορώ να δω τι γίνεται ακριβώς. Ένταξη ψηφοφορίας. Πέρας. Ήταν οριακό το αποτέλεσμα. 31 υπέρ, 29 κατά, μία αποχή. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 365 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αγκρή 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 367 υπέρ κατά να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την 367 υπέρ. Για την 367 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 367. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Α, ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 20 ψήφοι υπέρ, 39 κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν. Και τώρα περνάμε στην 113 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 369 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται ταυτόσημες οι 370 και καταπίπτει η 49. Και περνάμε τώρα στην επόμενη σελίδα. 373 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 έχει αποσυρθεί. 371 και 372. Α, όχι. Έχουν καταπέσει επίσης. Αγκρή 53 και 374. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 και ΙΜΚΟ 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 και 376 Είναι δύο διαφορετικές. Μία έχει συγγήτρια υπέρ και μία κατά. Να σας ψηφίσουμε μπροστά. 120 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και άλλη καταπίπτει φαντάζομαι. Το 375 κατέψει. Ήμκο 52. Επίση κατέψε 121. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ακριβώ 55. Was denn? So, 56. 56. Άγκρι 56. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε την 122 ελέγχουμε ηλεκτρονικά Πέρας πληροφορίες. Ναι, 36 υπέρ, 26 κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα. Ενοποιημένες τροπολογίες 6 και 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε αν θέλετε. Ευχαρίστως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 35 ψήφοι υπέρ και 26 κατά. Είναι κρίθη λοιπόν. Και περνάμε τώρα στη σελίδα 28. 392 και 394. Ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 396. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη σελίδα. 400, τροπολογία 400, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σελίδα 32. Τροπολογία 127. Πέμπτο τμήμα. Α, έχει αποσυρθεί. Άρα θα ψηφίσουμε σελίδα 32 την τροπολογία 407 έκτο τμήμα της κυρίας Ζόμερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 403 πέμπτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το επόμενο καταπίπτει. 407 έβδομο τμήμα και 405 πέμπτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Σελίδα 33, 411, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 130, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 131, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 61, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 414 υπέρ. Κατά. Αποχές κρίνεται. Να ελέγξουμε την 414. 414 ελέγχουμε. Beendet. πληροφορία. πληροφορίας. 38 υπέρ και 25 κατά. Σαφής. Consolidated Amendment 8, Ενοποιημένη 8. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Ήθελα να προσθέσουμε το soft στα soft drinks, όπου έχετε τον κατάλογο κατηγοριών. Εκεί που λέει drinks, να προσθέσουμε τη λέξη soft drinks. Ωραία, με την προφορική αυτή τροπολογία ψηφίσουμε την ενοποιημένη 8, υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Άρχεται η πληροφορία. Ένας από το ΕΛΚ περισσότερος από ό,τι πρέπει. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Απέριπτε, απερίφθη. Περνάμε λοιπόν στη συνέχεια. Τυπικά ψηφίσαμε για την προφορική τροπολογία και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την ενοποιημένη 8 ηλεκτρονικά. ηλεκτρονικά. Ist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 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 417. Α, όχι, έχει καταπέσει. 415 στη σελίδα 34. Ποιος είναι υπέρ 415. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 420 έχει αποσυρθεί. 437. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 67. 134 για τον 432. Υπέρ. Κατά. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να ψηφίσουμε. Άκρη 67, 134, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Την τροπολογία αυτή θα έπρεπε να την έχουμε ψηφίσει από μόνη της, γιατί δεν είναι τελείως ταυτόσιμη, ήταν σχεδόν ταυτόσιμη και γι' αυτό ε, δεν σήκωσε κανείς το χέρι του, γιατί έχουμε τρεις παρατηρήσεις για τρεις τροπολογίες. Ωραία, να τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Άγκρι 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές και αυτή απορρίπτεται. 432 υπέρ. Κατά. Και αυτή απορρίπτεται, αλλά αν θέλετε το ελέγχουμε για την 432 παρακαλώ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Και αυτή απορρίπτεται. Ωραία. 4.39. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4.30. Α, συγγνώμη, 439 έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 439. Περισσεύει ένας από το έλικα. Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ 30 κατά, δύο αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε φτάσει στην 4.30. 4.30. Να ψηφίσουμε και την 431, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.30. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ίνκο 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.36. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.35-4.27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.34 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 429 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 438 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ε, θεωρώ ότι εγκρίθηκε, αλλά στο ελέγξουμε για την 438, παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα ψηφορίας. 17 υπέρ και 44 κατά. Αχα, απερίφθη λοιπόν. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 440 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 441, 442 και ΙΜΚΟ 64. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ενοποιημένη υπαριθμό 9. Για την ε, υπέρ παρακαλώ, για την ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 9. Κατά. Απορρίπτεται. Αλλά ας το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. Ένα ψηφοφορίας. πέρας. «25 ψήφοι υπέρ, 36 κατά, μία αποχή απορρίπτεται». Και να περάσουμε στις τρεις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε κατά τμήματα, 137, 443 και 446. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα το πρώτο τμήμα Υπέρ παρακαλώ για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 453 weiter, Seite 39. Das ist mit 447. Bitte? Das ist mit 447. Second part of Splitwell Falls. Wir sind Seite 39. Βρισκόμαστε στη σελίδα 39. 453 είναι η τροπολογία. Τροπολογία 453 στη σελίδα 39. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 138 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 452 πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές. εγκρίνεται 454 πρώτο τμήμα και ΙΜΚΟ 68 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Abstimmung beendet. Ja, Das war knapp. 31 υπέρ και 29 κατά. Δύο εποχές. Υπέρ. κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Η Άλντα έχει ένα περισσότερο από ό,τι πρέπει τώρα. okay. Also. Λοιπόν. 31 υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται δηλαδή. Ωραία. 454 δεύτερο τμήμα και ΙΜΚΟ 68 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίες. ψηφοφορία. 28 υπέρ, 34 κατά. Απερίφθη λοιπόν. Εκατόν τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές, απερίφθη. Να ελέγξουμε. 138 τέταρτο τμήμα. Άρχιτε ψηφοφορία. Απερίφθη. Μικρή διαφορά, αλλά απερίφθη. Έχω καλά μάτια. 452 τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 τέτα, πέμπτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε και αυτό. Πέμπτο τμήμα 38. Πέρας. Επερίφθη. Άγκρι 69. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 451 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 455 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 452 τέταρτο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται. 454 τρίτο τμήμα υπέρ. 454 τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Ήμκο 68 τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται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 η γραμματεία μου λέει ότι μια απορρίπτει η 9, δεν μπορεί και η 10 να θεωρηθεί, η 10 ενοποιημένη τροπολογία να ψηφιστεί και πρέπει να τις ψηφίσουμε μεμονωμένα. Λοιπόν, 459, κράμερ υπέρ. 459, κράμερ υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Αγκρή 70, υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 464 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 464 έλεγχος. Abstimmung beendet. Πέρασε ψηφοφορίες. 30 υπέρ, 31 κατά ψήφι. 461 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 458. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 463. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ωραία, να ελέγξουμε. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρασε τη Ναι, άκουσε τον κόπο. 30 υπέρ, 32 κατά. Απερίφθη. 460 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 462 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία, να ελέγξουμε. Για την 462. Το έλκα έχει έναν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Τώρα μας εντάξει. Λοιπόν, 34 υπέρ, 27 κατά. Τώρα εγώ και κέρδισα όμως. Το είχα πει σωστά πριν. <laughs> 140. Κυρία Σόμερ. Ε, αυτή η τροπολογία που ψήφισαμε το 462 καταπίπτει λέγεται αν έχουν γίνει δεκτές όλες τις άλλες τροπολογίες που αναφέρον, προαναφέρονται και δεν ξέρω ελέξατε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ελέγξαμε, το ελέγξαμε. Ψηφίσαμε κιόλα. Και υπήρχε και πλειοψηφία υπέρ. Είμαστε στην 140. Υπέρ τη 140. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά βλέπω αρχίσετε και κουράζεστε. Από ό,τι κατάλαβα απερίφθη πάντως. Να ελέγξουμε 140. 140. EVP eine zu viel. Immer noch, jetzt. Το ΕΛΚ έχει ένα περισσότερος, τώρα εντάξει. Ω, oh, 44 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 467 είναι η επόμενη. Υπέρ. 467. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν σαράντα ένα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Wen habe ich denn abgelehnt? Nicht 470, 500. 470, 575. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 142. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 457 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Ωραία. Και η επόμενη καταπίπτει. 475 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 475. Πέρασε τις ψηφοφορίες. 29 υπέρ, 32 κατά. Ναι, απερίφθη πράγματι. Τώρα, 142, 456 και ΙΜΚΟ 70 ταυτόσημες υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται 457 και 473 ταυτόσημες. α, κατέπεσαν και περνάμε στην 471, 474 και 472 και αγκρή 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται άγκρι 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 457 και 476 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Ήμκο 71, υπέρ. Α, όχι, κατέπεσε. 143, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 477, υπέρ. Υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Τις 477 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα είναι, 457 και ήμικο 72. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Α... 144 και 457. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Immer noch. Jetzt. Απορρίπτεται 29 ψήφοι υπέρ, 32 κατά. 456. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Για την άκρη 74 παρακαλώ. so Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. 27 υπέρ 33 κατά. Και τώρα περνάμε στην 145 υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. 478 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Περισσεύει πάλι ένας από το ΕΛΚ. Πέρασε. Jetzt Σαφές το αποτέλεσμα. 35 η υπέρ, 24 κατά εγκρίνεται. 456. 456 υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία παριθμών 11. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ένταξη ψηφοφορίας. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Εξακολουθεί να περισσεύει. Τώρα εντάξει. Απορρίπτεται. 30 ψήφοι υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. Also, 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. άκρη 76 και 483. Ταυτόσημη υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 481 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 485 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 486 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Σελίδα 47, ΙΜΚΟ 73, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 78, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 74, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε για την 150 πρώτο τμήμα. Ένταξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Εντάξει με το ΕΛΚ. Εγκρίνεται. 32 ψήφοι υπέρ, 28 κατά. Και συνεχίζουμε στην 491 άγκρι 79 και 492. Α, αποσύρθηκε. Όχι, εντάξει, οι δύο πρώτες τότε. Υπέρ. Στη σελίδα 47 κάτω-κάτω είμαστε. 491 και άγκρι 79. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε στη σελίδα 48, 150 και άγκρι 80 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Έναξη ψηφορίας. Πέρας. 32 ψήφοι πέρ 28 κατά, εγκρίνεται. Άγκρι 81, ΙΜΚΟ 76. 4,93 και 4,94 υπέρ. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 κάτω κάτω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 497. Στη σελίδα 49, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 498. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 500. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 499 υπέρ. Κατά. Πρέπει να το ελέγξουμε, δεν το βλέπω. Γιατί την 499 παρακαλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφορίας. Beendet. Πέρας απορρίπτεται. 25 ψήφοι υπέρ, 33 κατά. Και περνάμε ταυτόσημες οι 151 και 501 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, ναι. Σε τμήματα, άγρι 83, και ΙΜΚΟ 77 σε 10 τμήματα. Θα γελάσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτονται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας για το τρίτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίθηκε. 31 ψήφοι υπέρ. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Καλά. Αποχές απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έκτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Έβδομο τμήμα υπέρ. κατά αποχές να το ελέγξουμε καλύτερα για το 7ο τμήμα παρακαλώ Bandits. Πέρας. Απορρίπτεται. 8ο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε για το 8ο τμήμα. Πέρας. Καλά το είδατε, απορρίπτεται. 32 κατά 29 υπέρ. Και περνάμε στο 1ο τμήμα υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Δέκατο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό απορρίπτεται. 502 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλλά αν να το ελέγξουμε, Μα θέλετε, για την 152. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 503. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε και αυτό γιατί είναι πολύ ωριακό το αποτέλεσμα. Για την 503 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 38 η ψήφη υπέρ. Εγκρίνεται. 504 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πεντακόσια επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 508 υπέρ. κατά αποχές να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 508 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 509 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 154. Μόνο την 154 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 511. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 155. Beendet. Πέρας. Απορρίπτεται. 514. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 515. Ακαταπίπτει. Και συνεχίζουμε στη σελίδα 52 με την 512. 512, δεύτερο τμήμα παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην 516. και 513 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 517. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 514. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. 514. δεύτερο τμήμα. Beendet. Πέρας και εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ 27 κατά. 518. Καταπίπτει. 514 και αυτή καταπίπτει. Ψηφίζουμε 514 τρίτο τμήμα Γκλένις Βίλμοντ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 519 Καταπίπτει, είπε τα 19. 5-13 και αυτή καταπίπτει. 156 στη σελίδα 53. Υπέρ. 156 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5-20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 5.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 84. Ήμκο 78 και 160 σε τέσσερα τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό απορρίπτεται. Και έτσι περνάμε στην 523 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 524 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο για την 524, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Na gut, da habe ich mich verschaut. Also das. Äh, Έκανα λάθος. Ναι, ήταν δικό μου λάθος, συγγνώμη. 47 η ψήφη υπέρ, εγκρίνεται. Εκατόν Υπέρ. Κατά. αποχές να το ελέγξουμε για την 161. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Ακόμα. Εντάξει. Εγκρίνεται. 32 ψήφοι υπέρ, 29 κατά. Και περνάμε στην 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε για την 162. Πάλι ένας περισσεύει από το ΕΛΚΑ. Μα βγάλτε έναν εκτός. Εγκρίνεται. 163. 163. Υπέρ. γιατί είναι 163. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 85. Υπέρ. Άγκρι 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 5.26. Δεν ε, ήταν παραδεκτή και περνάμε στην ΙΜΚΟ 79. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5.28 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 5.29 δεύτερο τμήμα. Σνέλχαρτ, υπέρ. Κατά. άποχες να το ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα της 529. Beendet. Πέρας. Abgelehnt. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην 530. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται, θεωρώ. Αλλά δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας και προβληματίζομαι. Να ελέγξουμε λοιπόν για την 530. Abstimmung beendet. Πέρας. Εγκρίνεται, εντάξει. Και περνάμε στη σελίδα 56. 531 πρωτοτμήμα. Υπέρ. Chris Davis. Υπέρ λοιπόν. Για την 531 πρωτοτμήμα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 531 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε για την 166 πρώτο τμήμα. Έλεγχος. Περισσεύει ένας από το έλκα Δικαίως ε, μπερδευτικά. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Και περνάμε τώρα στην άγκρη 87 υπέρ. Α, ξέχασα μία τροπολογία για να γυρίσουμε πίσω. Στην 166 παρακαλώ τρίτο τμήμα. Πρέπει να ψηφίσουμε και το τρίτο τμήμα της 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην άγκρη 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μήπως βιάζομαι, μήπως πάω γρήγορα. 166 τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 δεύτερο τμήμα υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 166 πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 αποσύρθηκε άγκρι 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έχουμε μια γλωσσική εισφύσεως και περνάμε στην 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι φιλελεύθεροι δεν ψήφισαν καθόλου. Σελίδα 57. 168. Λένε το υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται 168 πέρασε τις ψηφοφορίες 31 προς 30 ψήφους Αγκρή 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αγκρί 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 533 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αγκρί 96 και 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αγκρή 97 και 535 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 534 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 173 και 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 και 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 175 και 100 υπέρ

176 λέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άκρη. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχος. Πέρας. 30 υπέρ και 22 κατά. 9 αποχές. Εγκρίνεται. 536 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 537 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 538 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 540 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 541 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 542 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πολύ ωραία πάμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. 543 και ΙΜΚΟ 83. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ήμκο 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αγκρή 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 544 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 545 με μία προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Να ελέγξουμε την 545. Πέρας. Απορρίφθη. Και τώρα την 545 χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. ΥΜΚΟ 85. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 85 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 103 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 185, Αγκρή 105 και Ήμχο 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 551. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 546. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 547 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 549 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 550 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε 555. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 550, συγγνώμη, 550. Πέρασε ψηφοφορίες. Ναι, σαφέστα. Ε, 36 προς 25. 186. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτα. Ήμκο 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. ΥΜΚΟ 86. Beendet. Ναι, υπέρ, ξεκάθαρα υπέρ. 187 και ΥΜΚΟ 88, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Αγκρή 104, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρια 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρια 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 553 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 552 και αγκρία 108 Ταυτόσιμες. υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι 190 επισήρθη 554 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 555 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 556 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αγκρή 109, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται μάλλον, αλλά να ελέγξουμε. Αγκρή 109. So. Beendet. Πέρασε. Α, περίφθη. Ναι. 191. Γλωσσική είναι αυτή. Πρέπει να ψηφίσουμε. Α, 191. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η κυρία Έρμπερ έχει μια προφορική τροπολογία για την 110 για την Αγκρία 110, κυρία Βασκέρβερ. Ναι. Και για την 557. Η Αγκρία 110 και η 557 είναι τα αυτόσημες. Πρώτη κατάλληλη σήμανση των τροφίμων. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει εδώ ένας κατάλογος παραδειγμάτων που λέει ο, ο ακόλουθος κατάλογος συμπεριλαμβάνει παραδείγματα. Η Σκιώδης και η ίδια η ήταν σύμφωνοι να σημαίνονται ειδικά αυτά τα παραποιημένα, τα, τις απομιμήσεις των τροφίμων. Ωραία. Θα ψηφίσουμε την Αγκρία 110 με αυτή την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η ίδια προφορική τροπολογία για την 557 ή εντάξει. Α, όχι εντάξει. Ωραία. Ψηφίσουμε τώρα την 557 και την ΙΜΚΟ 89. Α, όχι, κατέπεσαν. Ναι, ναι, ναι, κατέπεσαν. ΙΜΚΟ 90. Δαφύρ. ΙΜΚΟ 90, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αγκρή 111 και ΙΜΚΟ 91, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. ΥΜΚΟ 91 δεύτερο τμήμα και άγρια 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. ΥΜΚΟ 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 558 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5... Όχι. 559 καταπίπτει. 193 με μια προφορική τροπολογία. Α, και αυτή καταπίπτει. Ωραία. 560. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 561 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 562 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Να ελέγξουμε την 562. beendet. Πέρασε. Απορρίπτεται. 27 προς 33. 563. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Περίφημα. Αλλά να ελέγξουμε αν θέλετε. 563 έλεγχος. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Όχι, ανακρίθη. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. 564, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 565 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 194 και 565 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 567 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 195 και Άγκρη 114 και Ήμκο 93. Α, η 195 έχει αποσυρθεί όμως. Λοιπόν, Άγκρη 114 και Ήμκο 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχος. Πέρας. Εγκρίνονται. Πεντακόσια Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. です。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 Δεν ξέρω ακριβώ γιατί, πάντως είχε γίνει δεκτό το 196. Μου λέει η γραμματεία. Και τη δίνω εμπιστοσύνη ναι. Λοιπόν, 198 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Άγκρα 115 και ΕΜΚΟ 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 569 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 573 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άκρη 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 570 πρώτο τμήμα και 199 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 570 δεύτερο τμήμα και 199 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 573 το τμήμα και 199 τρίτο τμήμα. Και το δεύτερο έχει αποσυρθεί μας. Λοιπόν, 573 τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άκρη 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 572 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άκρη 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 572 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άκρη 120 και 572 τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτα. Άκρη 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτα. 572 τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 570 τέταρτο τμήμα και 199 τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 571 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200 και 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 201 Υπέρ. Α, 200... Δεν είναι σωστός ο κατάλογος εδώ. Λοιπόν, 201. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε 201. Πέρας. Ναι, ναι, είναι κρίθη, ξεκάθαρα. Και τώρα, χτώσιμες ΙΜΚΟ 96 και ΑΓΡΕ 122. Όχι. Καταπίπτουν γιατί είναι κρίθη 21. 274 πρέπει να ψηφίσουμε για να δούμε. Όχι. Σε θεολογικέ σκέψει περνάμε τώρα. Ένα. Ένα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Σόμερ. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τρία, Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ακρί 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ακρί 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 και αγκρί 3. Το πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. επτά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται άγκρη 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Σελίδα 67, στην 12 και άγρι 6, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 202, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 203, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206, συγγνώμη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Στη 18 λοιπόν, σελίδα 68, υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Γιατί 18 παρακαλώ να ελέγξουμε. Ε; Πέρας. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209 και 210 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 213, 214 και 217 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε λοιπόν άμα θέλετε. 213, 216, 217 να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. 22 προς 39. Μία αποχή. Απορρίπτεται. Άγκρι 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 218 Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 222. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 222. Check beendet. Με μεγάλη διαφορά απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 221. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 21. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 223. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην άγκρη 13 και στην 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 23 στην 23 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 230 και ημκο 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 236 κάτω στη σελίδα 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. εγκρίνεται, συγγνώμη. Να το ελέγξουμε, αν θέλετε, για την 27 έναρξη ψηφοφορίας. Abstimmung Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 2.37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη 237 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Εντάξει. 2.38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Για την 2.38. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29 προς 28 ψήφι. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 2.39. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 241 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην επόμενη σελίδα περνάμε τώρα. Άγκρι 15. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 245 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνήθως έχω δίκιο, αλλά όχι πάντα φυσικά. Και περνάμε στα 32 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 16. Κατά. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 14. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόεδρε, να παρακαλέσω πριν την τελική ψηφοφορία να κάνουμε μια τελική, ένα διάλειμμα για να μπορέσω να διαβουλευτώ λίγο με την ομάδα μου. Όντω, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα μικρό διάλειμμα. Λέω 12 και 1. 12 και 10. Ένα διάλειμμα μέχρι τις 12 και 10. Άντε, 12 και 4. 12 και 4. 15 λεπτά διάλειμμα, λέει ο Πρόεδρος.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 liebe Kolleginnen und Kollegen, dear friends, 15 minutes are over. Συνάδελφοι, πέρασαν 15 λεπτά. A big, uh, big compliment to all members. Να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, πήγε εξαιρετικά η ψηφοφορία. Δύο ώρες και 40 λεπτά. Περάσαμε γρήγορα γρήγορα 900 τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Οι πολιτικές ομάδες ε, διαβουλεύτηκαν και τώρα ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας, της τελικής ψηφοφορίας, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά. Πρώτη ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης στο σύνολό της. Ε, έναρξη ψηφοφορίας sagst, wir sollen das The vote is closed. Ένας ψηφοφορίας. Και 51 οι ψήφοι υπέρ, 4 η ψήφοι κατά, 5 αποχές. Και να ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο νομοθετικής πρότασης ε, και πάλι ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Abstimmung Πέρας. 52 οι ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια να συγχαρούμε την κυρία Ζόμερ και για την έκθεση και για όλη τη δουλειά που έκανε. Συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Και διακόπτουμε για σήμερα. Συνεχίζουμε στις 3 με τις υπόλοιπες ψηφοφορίες. Καλή όρεξη και τα λέμε το απόγευμα.